το σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι η παρουσίαση της έκθεσης, ετήσιας έκθεσης του ελεκτικού συνεδρίου για το έτος 2009. Θα μας παρουσιάσει την έκθεση ο πρόεδρος του ελεκτικού συνεδρίου, ο κύριος Βίκτορ Μανουέλ Ντασίλβα Καλντέρα. Έχετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητά μελή, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη τιμή για μένα να πάρω μέρος της συνάντησης αυτή σήμερα για την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εφαρμογή του προϋπολογισμού του 2009. Την έκθεση σας παρουσίασα ήδη σε εσά κύριε Πρόεδρε και στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου. Θα ήθελα να σας μεταφέρω τέσσερα βασικά μηνύματα που περιλαμβάνονται στην έκθεση. Πρώτον, οι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίδουν μια γνήσια παρουσίαση, μια δίκαιη και γνήσια παρουσίαση των δημοσιονομικών και των αποτελεσμάτων των οικονομικών επιχειρήσεων όπως επίσης και των ε, ροών των οικονομικών. Είναι η τρίτη χρονιά όπου οι λογαριασμοί συνολικά θεωρούνται ότι είναι ακριβείς και αξιόπιστοι. Σχετικά με την νομιμότητα και την κανονικότητα, το ελεγκτικό συνέδριο εκφράζεται ελεύθερα και στον τομέα των εσόδων και στον τομέα των υποχρεώσεων, όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Όμως, και αυτό είναι το δεύτερο μήνυμα, οι πληρωμές από τον προϋπολογισμό επηρεάζονται από λάθη, εκτός από δύο τομείς των δαπανών. Οι δύο εξαιρέσεις είναι οι διοικητικές δαπάνες και οι οικονομικές και, και χρηματοπιστωτικές υποθέσεις. Σε όλους τους άλλους τομείς υπάρχουν συγκεκριμένα επίπεδα λαθών. Θα συγκεντρώσω την προσοχή μου σε δύο τομείς όπου υπάρχουν τέτοιες δαπάνες, στη γεωργία και στη συνοχή. Στη γεωργία και στους φυσικούς πόρους το επίπεδο ε, λάθους είναι υψηλότερο από το 2008 Παρ' όλα αυτά τα αποτελέσματα είναι συμβατά με τις εκτιμήσεις που έχει κάνει το ελεγκτικό συνέδριο ότι τα συστήματα που χρησιμοποιούνται είναι μόνο επιμέρους αποτελεσματικά. Συστήνουμε τη μείωση των επιπέδων λαθών μέσω της βελτίωσης των συλλαγωμένων πληροφοριών και δεδομένων βάσεων έτσι ώστε να εφαρμοστούν σωστότερα οι κανόνες σχετικά με την συντήρηση και τη χρήση της γης. Στον τομέα της συνοχής, ε, και εδώ έχουμε να κάνουμε με το 1 τρίτο του προϋπολογισμού, η κατάσταση παραμένει όπως και στο παρελθόν. Το ποσοστό λάθους είναι άνω του 5%. Τα περισσότερα λάθη τα οποία έχουν βρεθεί ε, οφείλονται στις αδυναμίες των εθνικών αρχών να εφαρμόσουν τους κανόνες σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την επιστροφή των αχρεωστήτων ε, πληρωμένων ποσών πάρα πολλά λάθη θα έπρεπε να έχουν διορθωθεί από τα κράτη-μέλη πριν ε, καταστήσουν έγκυρες δαπάνες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ακριβώς έχει δείξει ο έλεγχος που έχουμε κάνει. Αν συγκρίνουμε τα αποτελέσματα με τον προηγούμενο χρόνο, βλέπουμε ότι πολύ σημαντικές αλλαγές έχουμε στον τομέα της συνοχής. Και έρχομαι τώρα στο τρίτο μήνυμα. Έχουμε μικρότερα επίπεδα βέβαια λαθών από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια και στο σύνολο του προϋπολογισμού το επίπεδο λαθών έχει κατέβει γενικότερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Παρ' όλα αυτά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην ορίσουμε συγκεκριμένους τρόπους πορείας των δημοσιονομικών και νομίζω ότι ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες ε, μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια το 9 δεν ήταν πολύ διαφορετικό από το 8. Παρ' όλα αυτά η μείωση του επίπεδου των λαθών τα, που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια θα συνεχιστεί εφόσον τα συστήματα ε, είναι αποτελεσματικά αλλά όχι συνολικά αποτελεσματικά και έρχομαι στο τελευταίο αν θέλετε κεντρικό μήνυμα οι πληροφορίες τις οποίες δίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις ανακτήσεις ποσών δεν είναι απόλυτα αξιόπιστες και δεν μπορούν ε, επί της ουσίας να συγκριθούν με τα επίπεδα λαθών τα οποία υπολογίζει κατά προσέγγιση το ε, ελεγκτικό συνέδριο. Υπάρχουν αρκετές πρωτοβουλίες τις οποίες πρέπει να αναλάβουμε σχετικά με την βελτίωση της ε, δημοσιονομικής διαχείρισης της Ένωσης μακροπρόθεσμα η ετήσια μας έκθεση φέτος επιβεβαιεί τα αποτελέσματα και τις συστάσεις τις οποίες έχουμε ήδη δηλώσει ε, στο παρελθόν σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Η βελτίωση της ποιότητας των δαπανών είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Η απλοποίηση των νομοθετικών πλαισίων και πιο οικονομικά ε, συστήματα ελέγχου για τη μείωση του επίπεδου των λαθών θα συνεισφέρουν προς την κατεύθυνση αυτή. Νωρίτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια πρόταση αναδιατύπωσης του δημοσιονομικού κανονισμού ε, σχετικά με αυτή την δήλωση. Το ελεγκτικό συνέδριο θεωρεί ότι περιλαμβάνει ορισμένες προτάσεις θετικές για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα οδηγήσουν στη βελτίωση της διαφάνειας. Η απλοποίηση τομεακών νομοθετικών όμως δημάτων παραμένει ένα πολύ σημαντικό ε, εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί για να βελτιωθεί η ποιότητα των δαπανών. Τον επόμενο χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει νομοθετικά προγράμματα για διαφορετικές πολιτικές για την επόμενη προγραμματική περίοδο στον τομέα των δαπανών. Όταν υπάρχουν αναθεωρήσεις των προγραμμάτων δαπανών, το Ελεκτικό συνέδριο προτείνει την εφαρμογή ορισμένων αρχών έτσι ώστε η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία να είναι σαφής, οι στόχοι να είναι σαφείς επίσης τα προγράμματα να είναι ρεαλιστικά και απλά όσο τουλάχιστον αυτό είναι ευθέτως δυνατό και να υπάρχει ξεκάθαρη δυνατότητα ορισμού υπολόγων. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, θα πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να δαπανώνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη για όλους και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που κάνει προτάσεις νομοθετικές και εφαρμόζει τον προϋπολογισμό και για τα κρατημέλη γιατί διαχειρίζονται σε καθημερινή βάση το 80% του προϋπολογισμού αυτού αλλά και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σαν συνομοθέτες όπως επίσης και στο ελεγκτικό συνέδριο που είναι ο εξωτερικός σας ελεγκτής. Το ελεγκτικό συνέδριο λοιπόν θα κάνει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε τα κοινοτικά χρήματα να δαπανώνται σωστά. Σα Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρους τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ακούσουμε τώρα τον Επίτροπο Αλγκίντρας Σεμέτα. Έχετε το λόγο κύριε Επίτροπε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε Καλντέρα, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, και εξότιμα μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου. Πριν από δύο μέρες, ο πρόεδρος Καλτέρα και εγώ ήδη είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και να συζητήσουμε την ετήσια έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου με τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να επισημάνω εδώ τα βασικά στοιχεία της συζήτησης και τα πρωταρχικά μας συμπεράσματα. Πριν επισέλθω στο κυρίως θέμα, θα ήθελα να επισημάνω τον επικοδομητικό διάλογο που είχε το ελεκτικό συνέδριο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ελεγκτής και ο ελεγχόμενος δηλαδή, και να ευχαριστήσω για την αγαστή αυτή συνεργασία τον πρόεδρο Καλντέρα. Χαίρομαι με την αναγνώριση της πρόοδου που έκανε το ελεκτικό συνέδριο. Και είναι πολλά τα θετικά μηνύματα της ε, ετήσιας έκθεσης. Βλέπω βέβαια και κάποιες ε, επικρίσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να παρακολουθήσει εκ του και να εφαρμόσει τις συστάσεις του ελεκτικού συνεδρίου. Τα βασικά μηνύματα της έκθεσης του ελεκτικού συνεδρίου θα καθοδηγήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανάληψη της υποχρέωσής της για την διαχείριση του προϋπολογισμού. Για τρίτη συνεχή χρονιά είχαμε μια θετική ε, γνώμη του ελεκτικού συνεδρίου και θεωρήθηκε ότι οι λογαριασμοί χωρίς επιφύλαξη δίνουν μια αληθή και ακριβωδική εικόνα της κατάστασης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα αυτό γιατί αποδεικνύει τα ε, θετικά αποτελέσματα της λογιστικής μας μεταρρύθμισης. Βέβαια το ελεκτικό συνέδριο επισημαίνει κάποιες αδυναμίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει αυτές τις αδυναμίες που επισημαίνονται και να συνεχίσει την βελτίωση των λογιστικών της πρακτικών. Σε ό,τι αφορά την νομιμότητα και τον θεμητό χαρακτήρα των διαφόρων συναλλαγών, χαίρομαι γιατί μειώθηκε το γενικό ε, επίπεδο λάθους και τα έσοδα και η αναλήψη υποχρεώσεων είναι ε, νομότυπες σε όλες τις περιπτώσεις και 90% των πληρωμών που έγιναν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό είναι απαλλαγμένες από οποιοδήποτε λάθος. Αυτή η αναγνώριση είναι ένα θετικό μήνυμα ότι οι προσπάθειές μας να βελτιώσουμε τον έλεγχο αποφέρουν καρπούς. Και αυτό ε, επιτεύχθη χάρη σε μια σημαντική μείωση του ποσοστού λάθους ε, στη συνοχή χάρη στην, στο διευρυμένο εποπτικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με εκ των προτέρων ε, αξιολογήσεις των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών. Επίσης, ε, ε, οφείλονται στην αυστηρή μας ε, προσέγγιση σε ό,τι αφορά την καταβολή των πληρωμών, ακόμη και την αναστολή του σε περίπτωση που εντοπίζονται προβλήματα. Επίση, το ελεκτικό συνέδριο αναγνωρίζει την υψηλή ποιότητα των πληροφοριών για τι ανακτήσει ποσών που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αύξηση της αξίας των κονδυλίων που ανακτώνται από σχέδια τα οποία ήταν ελαττωματικά ή πέστηκαν λάθη είναι επίσης ενδεικτικό της αποφασιστικότητας για χρηστή διαχείριση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το λεκτικό συνέδριο επισημαίνει προβληματικές ε, εκθέσεις εκ μέρους των κρατών μελών και αυτή η κατάσταση πρέπει να διορθωθεί και για τα επιστάμενα προγράμματα αλλά και για την επόμενη γενιά προγραμμάτων που υπόκειται σε κοινή διαχείριση. Φυσικά συμμερίζομαι την επιφυλακτικότητα του Πρόεδρου Καλντέρα όταν ε, μιλά για πιθανές διακοιμάνσεις του ποσοστού λάθους, ιδιαίτερα στο μέλλον ε, για τη συνοχή. Επίσης, συμφωνώ με το λεκτικό συνέδριο που επισημαίνει κάποιες αδυναμίες στα συστήματα κρατών μελών και κάποια άλλα επιμέρους θέματα της κοινή διαχείρισης. Κατά τη γνώμη μου, στο μέλλον θα πρέπει να έχουμε ελεκτικούς μηχανισμούς που θα είναι αποδοτικοί, θα πρέπει να προστατεύσουμε τους, κανόνε τους κανόνες επιλεξιμότητας, να μειώσουμε το λάθος και να βελτιώσουμε την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τις χρηματοπιστωτικές διορθώσεις και τις ανακτήσεις ποσών. Βέβαια, ο κατάλογο αυτό για το βελτιώσεων δεν είναι εξαντλητικέ. Οι συζητήσει μα έδειξαν ότι υπάρχουν και άλλες προκλήσεις ενώπιόν μας. Για παράδειγμα, μεγαλύτερη λογοδοσία για του πιο σημαντικού χρηματοπιστωτικού φορεί, ιδιαίτερα στα κράτη-μέλη. Μία αποτελεσματική ε, πολιτική ελέγχου. Επίση, κατά την προ... προπαρασκευή του... της δημοσιονομικής μεταρρύθμισης, θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στον αντίκτυπο και όχι ε, στη, στο προηγούμενα στάδια. Και φυσικά θέλουμε σαφείς στόχους και δείκτες ε, απόδοσης και επίδοσης. Επίσης, ε, έχουμε το σχέδιο για την πολιτική καταπολέμηση απάτης μέχρι το 2014. Το πρόγραμμα αυτό επισημαίνει τους βασικούς στόχους και τα βήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να έχουμε και στο μέλλον θετικές δηλώσεις αξιοπιστίας του ελεκτικού συνεδρίου. Πάντως το πρόγραμμά μας θα είναι πολύ σημαντικό και για τις μελλοντικέ μας δράσεις. Είμαι γενικώ ικανοποιημένο γιατί η ετήσια έκθεση του 2009 αναγνωρίζει την αποδοτικότητα των προσπαθειών μας και επίση ε, θα συμβάλλει στον περαιτέρω προβληματισμό μας για την εξασφάλιση χρηστής ε, δημοσιονομικής διαχείρισης του κοινοτικού προπολογισμού στη φάση που προετοιμάζουμε και τη μελλοντική γενιά των προγραμμάτων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θα περάσουμε τώρα στον κατάλογο των αγοριτών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το λόγο έχει η κυρία Ίγκεμπορκ Κρέσλε. Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Ελεκτρικού Συνεδρίου, αγαπητοί επιτρόποι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα έχουμε μπροστά μια πολύ θετική μέρα, γιατί για πρώτη φορά μπορούμε να ε, υπολογίσουμε ότι η Επιτροπή Παρόζο θα περάσει το όριο, το όριο του 2% και γι' αυτό η έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου είναι ένα πολύ καλό μήνυμα, ιδίω για όλους όσους εργάστηκαν για το οικοδόμημα αυτό. Και βλέπουμε όταν η Κομισιόν ε, δράσει αποτελεσματικά, πετυχαίνει αποτελέσματα. Εξετάζουμε τώρα το αποτέλεσμα στις λεπτομέρειες. Ε, πολλά από αυτά εξαρτώνται από τον διακανονισμό. Είναι σωστό αυτό και προς τα εκεί θα πρέπει να κινηθούμε και στο μέλλον. Εάν η Κομισιόν ξεκινήσει να μεταρρυθμίσει τον κανονισμό για τις δημόσιες αγορές και τους δημόσιους διαγωνισμούς θα έχει πετύχει το μεγαλύτερο βήμα προς το εμπρός προς ε, θετικές δηλώσεις αξιοπιστίας. Προς όλους εκείνους που ισχυρίζονται ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός εκτίθεται σε σημαντικούς κινδύνους, έχω να πω ότι οπωσδήποτε τα ευρωπαϊκά χρήματα θα πρέπει να ελέγχονται με, ελέγχονται με μεγαλύτερο ε, μεγαλύτερη σοβαρότητα από ότι οι εθνικές δαπάνε. και το βλέπουμε αυτό πάντα όταν κινούμεθα στα κράτη-μέλη όπου βλέπουμε ότι καμιά φορά υπάρχουν οι εθνικοί κανόνε μόνο επειδή υπάρχουν ευρωπαϊκοί και γι' αυτό θα πρέπει να ενθαρρύνουμε και να καλέσουμε τα κράτη-μέλη να ελέγχουν τα εθνικά τους ε, ταμεία με τον ίδιο τρόπο όπω τα ευρωπαϊκά και τα ναύαλη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ελεκτρικό συνέδριο και να του πω ότι είμαι κάπως απογοητευμένη από την ετήσια έκθεση. Το είπα ήδη. Η ετήσια έκθεση έχει λιγότερες πληροφορίες από ό,τι στο παρελθόν. Χρειαζόμαστε στοιχεία για τα ποσοστά ασφάλματος. Τα είχαμε πάντα για τα ελευθερικά ταμεία, τώρα όχι. Κυρίε και κύριοι, δεν είμαστε στην πιαγωγή εδώ. Κοινοβούλιο είμαστε και εξωτόμεθα να έχουμε τα στοιχεία αυτά στα χέρια μας. Και όταν ε, θυμηθώ τις ακροάσεις των μελών του ελεκτικού συνεδρίου ε, θυμάμαι ότι μας υποσχέθηκαν να συνεργαστούν στενά με το Κοινοβούλιο και δεν το κάνουν μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, σας, σας ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος της Σοσιαλιστικής ε, και Δημοκρατικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Γιώργος Σταυρακάκης. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχήν να χαιρετήσω την ετήσια έκθεση και να συγχαρώ τον Πρόεδρο του Καλντέρα και όλα τα μέλη του Ελεκτρικού Συνεδρίου για το έργο του, Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστώ τον κύριο Ρουσέ για την στενή και πολύ θετική συνεργασία που είχαμε μαζί του. Ο ρόλο μα ω Κοινοβούλιο είναι η λογοδοσία προ του πολίτε. Πρέπει να είμαστε σίγουροι λοιπόν ότι τα χρήματα των φορολογουμένων χρησιμοποιούνται σωστά, με διαφάνεια και όπως πρέπει. Ελπίζω ότι η έκθεση για τις εξωτερικές υπηρεσίες που θα υποβληθεί αργότερα θα ακολουθεί στην ίδια γραμμή που είχαμε μέχρι τώρα, γιατί βελτιώνεται η κατάσταση, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά που θα πρέπει να γίνουν. Στην σημερινή οικονομική και κοινωνική κρίση, η επιτήρηση και ο έλεγχος των ε, οικονομικών είναι όσο πάει και πιο σημαντικό. και το Κοινοβούλιο μαζί με το Ελεκτικό Συνέδριο έχουμε αποφασίσει να λύσουμε τα προβλήματα για να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Τώρα σας ευχαριστώ. Ο Γιώργος Χατζημαρκάκης εξονόματος τη ομάδα του. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σαμέτα, Πρόεδρε Καλτέρα, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ελεκτικό Συνέδριο για την έκθεσή του. Οι εργασίε τη υπηρεσία σα, κύριε Καλντέρα, εξυπηρετούν θαυμάσια τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Αυτό που είναι καλό είναι ότι συνεχίσετε η θετική εξέλιξη στη μείωση του επίπεδου σφάλματο. Αυτό ξεκίνησε ήδη με τον Επίτροπο Κάλλα. Στην έξι σήμερα υπάρχουν βελτιώσει όσον αφορά την συνοχή, μικρές ε, επιδεινώσει όσον αφορά τη γεωργία. Παρ' όλα αυτά δεν πρέπει να επαναφτύσει τι ε, δάφνε τη Κομισιόν πιστεύουμε ότι η βελτίωση οφείλεται σε δειγματολογικούς ελέγχους. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ορμή που υπάρχει από την πρώτη απαλλαγή του προπολογισμού μετά τη της αγώνας για να μπορέσουμε να βελτούμε στο μέλλον. Θα ήθελα να σας πω ότι η φετινή ετήσια έκθεση του ελεκτικού συνεδριού είναι η 16η σε σειρά που δεν καταλήγει σε θετικό αποτέλεσμα σφαιρικά. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να αποφύγουμε τις ε, σπατάλες. Εγώ ως εισηγητής έχω να προτείνω τα εξή. Καταρχήν θα πρέπει να δράσει ακόμα πιο σκληρά η Κομισιόν όταν υπάρχουν σφάλματα. Πώς είναι δυνατόν 10 χρόνια μια ε, χώρα όπως η Ελλάδα δεν υπέστη καμία ε, κύρωση ενώ υπήρχαν αυτές οι ατασταλίες. Δεύτερον, όσον αφορά τα χρεωσίδως καταβληθέντα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, το ποσοστό επανάκτησης είναι 10%. Τα κράτη-μέλη δίνουν 50% από το εθνικό προπολογισμό το δικό τους και το 50% έχει από την κοινότητα. Θα ήθελα να σας πω, από το 1994, στον τομέα της πολιτικής συνοχής μέχρι το έτος 2006, τα κράτη-μέλη είχαν πάρει αχρεωστήτως 7,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι στοιχεία που τώρα είδαμε. Η το ποσοστό θα ήταν μόνο 709 εκατομμύρια. Βλέπετε λοιπόν το ποσοστό του 10%. Τα κράτη-μέλη δεν είναι σε θέση να κάνουν τους υπολογισμούς σωστά. Το είπε το ηλεκτρικό συνέδριο και γι' αυτό λέω θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να έχουν επιτέλους εθνικές δηλώσεις διαχείρισης που να υπογράφουν. Ταυτόχρονα η Κομισιόν θα πρέπει να αναλάβει πολιτικά την ευθύνη με την υπογραφή του Προέδρου Μπαρόσο τουλάχιστον κάτω από την συνθετή έκθεση των ετησίων δραστηριοτήτων. Θέλουμε όμω να έχουμε και μια έκθεση αξιολόγηση, όπω προέρχεται αυτή από τι αιτήσεις τη Αβώνης. Κυρίε και κύριοι, πολλά πρέπει να βελτιωθούν. Γενικά ευχαριστώ όμω τον Ευρωπαϊκό Συνόδιο για την έκθεσή του. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο Πράσινη. Συνάλφο Μπαρτ Στάε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όταν διάβασα την ετήσια έκθεση του ελληντικού Συνεδρίου είχα μια αίσθηση déjà vu. Είναι κάτι το οποίο διαβάζουμε κάθε χρόνο εδώ και πολλά χρόνια. Καταρχάς υπάρχουν πολλά συγκεκριμένα λάθη στον τομέα της συνοχής, στον τομέα της κοινή αγροτικής πολιτικής, στη βοήθεια για την ανάπτυξη και στην εκπαίδευση. Βλέπουμε ότι τα συστήματα ελέγχου δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά και δεν μπορούν να διορθώσουν ε, τα υπερβολικά κόστη τα οποία μερικές φορές διαπιστώνονται. Και είναι μερικές φορές επίσης δύσκολο για τα κράτη-μέλη να γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν. Μιλάμε τώρα για τομεί οι οποίοι μπορεί να καλύπτουν και το 80% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Το θέμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε θέση να συνδράμει τα κράτη-μέλη προς την κατεύθυνση αυτή. Συμφωνώ λοιπόν με τον Πρόεδρο του ελεγκτικού συνεδρίου που ε, απαιτεί να υπάρχουν δηλώσεις αξιοπιστίας οι οποίες να υπογράφονται από τον εκάστοτε υπεύθυνο υπουργό. Και προφανώς αυτό μπορεί να οδηγεί και στη λήψη ε, κυρώσεων. Κύριος Τσαρνιέσκη. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το ελεγκτικό συνέδριο είναι ένας σημαντικός ελεκτικός φορέας, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα είδος αστυνομικού, βέβαια φιλικός αστυνομικός, αλλά έχω την αίσθηση ότι μερικές φορές παρά είναι επίκης και μεγαλόψυχος αυτός ο αστυνομικός και ο ελεκτής απέναντι στον ελεγχόμενο. Τα συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης του ελεκτικού συνεδρίου είναι θετικά αλλά δεν είναι ιδεώδη αυτά τα συμπεράσματα. Έχω την αίσθηση ότι πολλοί άνθρωποι στην Ευρώπη θεωρούν, κρίνουν με πολύ ε, απεσιόδοξο τρόπο το έργο του ελεκτικού συνεδρίου. Το ελεκτικό συνέδριο θα πρέπει να είναι ένα πραγματικά αξιόπιστο ελεκτικό συνέδριο για να ανακτήσει το κύρος της Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στους πολίτες και τους φορολογουμένους. Για να είναι όμως αξιόπιστο το ελεκτικό συνέδριο θα πρέπει να είναι πολύ πιο σχολαστικό. Σήμερα το ελεκτικό συνέδριο μας είπε ότι χαιρόμαστε που κατά 95% το ποτήρι είναι πλήρες. Πιστεύω όμως ότι πολλοί φορολογούμενοι θα διαρωτηθούν. Γιατί κατά 5% αυτό το ποτήρι είναι άδειο. Πολλό δε μάλλον που σε μεγάλο βαθμό το ποτήρι αυτό είναι άδειο πάνω από 5%. Ο έλεγχο σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να είναι πολύ πιο διεξοδικό ε, από ό,τι γίνεται στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό θα ήθελα να ε, παροτρύνω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πιέσει τα κράτη-μέλη να επιστρέψουν τα κονδύλια που αχρεωστήτω έλαβαν. Ευχαριστώ. Εκ μέρου ε, τη ε, ΓΚΟΕ, Ενωμένη Αριστερά, το λόγο έχει ο Σερεν øh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε εδώ μια καλή έκθεση μπροστά μας. Ε, αυτό που βλέπουμε είναι ότι μειώθηκε ο αριθμός ε, ε, των σφαλμάτων. Ενώ λοιπόν, θα το εξελίξουμε αυτό. Το εξαρτάται από δύο πράγματα. Καταρχήν από το σημείο εκκίνησης και από την άλλη από τις προσδοκίες που έχουμε. Το σημείο εκκίνησης ήταν πάρα πολύ κακό. Δισεκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν αντικανονικά. Και γι' αυτό οι προσδοκίες ήταν να υπάρχουν βελτιώσεις αφενός και αφετέρου να υπάρχουν σημαντικές βελτιώσεις σε όλους τους τομείς. Και αυτό έγινε. Σε ορισμένου τομεί δεν υπάρχουν πια αχρεωστήτω κατευληθέντα ποσά. Από την άλλη μεριά, το επίπεδο των αχρεωστήτω κατευληθέντων είναι τεράστιο, απαράδεκτο. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα αυξήθηκε. Αυτό είναι απαράδεκτο. Στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, ο Επίτροπο Εμέτα πρόσφατα είπε αυτό που επανέλαβε και σήμερα, ότι το γενικό ποσοστό μείωση του σφάλματο ήταν το αποτέλεσμα τη δέσμευση τη Κομισιόν. Πολύ ωραία. Θαυμάσια. Ε, να πενέσω κι εγώ την ε, Εκτελεστική Επιτροπή γι' αυτό. Αλλά το θέμα είναι ποιος ήταν όμως υπεύθυνο για τα σφάλματα, ποιος θα είναι υπεύθυνο όταν επαναληφθούν τα σφάλματα αυτά του χρόνου. Μάρτα Η ε, κυρία Μάρτα Ανδρέασεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Τα τελευταία 16 χρόνια το ελεκτικό συνέδριο δεν έδινε απαλλαγή για μεγάλο τμήμα του προπολογισμού. Και αυτή τη αυτό το χρόνο δεν έχουμε καμία διαφορά. Μα μιλούν για σφάλματα. Το είδο όμω των ατασταλιών που ανακαλύπτει το ελεκτικό συνέδριο ξεπερνούν το χαρακτηρισμό του σφάλματο. Μία τέτοια κατάσταση θα προκαλούσε το κλείσιμο μια εταιρεία, τη χρεοκοπία τη στον ιδιωτικό τομέα και την παρέτηση ή μάλλον ε, απόλυση των διευθυντών. Δυστυχώ τα χρήματα των φορολογουμένων ε, ξοδεύτηκαν με ασφαλμένο τρόπο και τουλάχιστον 6 δισεκατομμύρια λίρες λίρε μας λέει το ελεκτικό συνέδριο ότι καταβλήθηκαν αχρεώστατα. Πού έγκυται το πρόβλημα? Στην έλλειψη ευθύνη, υπευθυνότητα και λογοδοσία. Βέβαια η Επιτροπή κατηγορεί τα κράτη-μέλη, αλλά η η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευθύνεται λόγω των ελαττωματικών ελέγχων για τα λάθη αυτά. Θα πρέπει να θεσπίσει κανόνες και να επιβάλλει κυρώσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη-μέλη που παραβιάζουν τις διατάξεις αυτές. Δυστυχώ αυτή την κατάσταση έχουμε κάθε χρόνο και παρόλα αυτά ζητούμε συνεχώ αύξηση του κοινοτικού προπολογισμού. Δεν υπάρχει καμία πια ελπίδα ότι ο Ευρωπαϊκό Προπολογισμό θα λάβει θετική ανεπιφύλακτη γνώμη από το ελεκτικό συνέδριο. Ο μοναδικό τρόπο για να προστατεύσουμε τα χρήματα των φορολογουμένων μα είναι να μειώσουμε δραστικά τον κοινοτικό προπολογισμό. Ο κύριος Κάμερον με την αποδοχή του 2,9% αύξηση για τον προϋπολογισμό του 2011 απέτυχε παταγωδός στο έργο του και οι Βρετανοί φορολογούμενοι ε, ζητούν ε, να διεκδικήσετε σημαντική μείωση του προϋπολογισμού του 2011 κύριε Κάμερον. Μην γεγραμμένο μέλος τώρα θα λάβει το λόγο ο κύριος Έρνχάουζερ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Ναι, είναι σωστό, το ποσοστό σφάλματο στο τομέα τη συνοχή μειώθηκε σημαντικά από το 2007 από 54% στο 36% το 2009. Είναι σωστό. Αυτά είναι στοιχεία που πρέπει και εγώ να αναγνωρίσω. Αλλά όπω είπε και ο ίδιο η εισηγητή, αν τα εξετάσουμε σε λεπτομέρειε τα στοιχεία αυτά και να δούμε από πού προέρχονται, θα πρέπει να τα ε, θέσουμε σε αναλογία με τα άλλα. Ε, ελέγχεται στην έκθεση του ηλεκτρικού συνεδρίου ότι τα συστήματα ελέγχου στον τομέα της συνοχής δεν είναι αποτελεσματικά και λέγεται ότι τουλάχιστον το 3% των χρημάτων αυτών δεν θα έπρεπε να έχουν καταβληθεί. Απέχουμε ακόμα πολύ, δηλαδή, ακόμα και για τον Επίτροπο Γιωάννησα να διορθώσει την κατάσταση αυτών των τομέα. Όσον αφορά την αύξηση του σφάλματος στον τομέα της Γεωργίας, πρόκειται για πιστοδρόμηση. Γιατί ταυτόχρονα έχουμε ε, έχουμε την περίπτωση στην οποία καταβάλλονται ποσά σε δισεκατομμυριούχους και δεν θεωρούνται εσφαλμένα, ε, εσφαλμένα καταβεβληθένα τα ποσά αυτά. Πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσον ξέρουμε ποιος θέλει για την καταβολή των χρημάτων αυτών, κατά πόσον τα χρήματα αυτά θα επιστραφούν και μου φαίνεται ότι είναι σημαντικό στο μέλλον το ηλεκτρικό συνέδριο να μην εξετάζει μόνο κατά πόσο ήταν σωστά κατεβλημένα τα χρήματα αυτά, αλλά και κατά πόσο χρησιμοποιήθηκαν σωστά. Η απουσία του κυρίου Οντή, ο κύριος Ιβάν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Καλντέρα, τον πρόεδρο Καλντέρα, για μια σαφέστατη και πλήρη έκθεση σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2009. Να διευκρινίσω εδώ κάτι το οποίο έχει αρκετά μεγάλη σημασία. Κάθε πέντε χρόνια εμείς εκλεγόμεθα και ο Ευρωπαίος Φορολογούμενος μας στέλνει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο οποίος μέσω της προστιθέμενης αξίας που προσφέρει μας δίνει τη δυνατότητα να, να δουλεύουμε εδώ. Ο προϋπολογισμός λοιπόν του 2009 δεν είναι ένας καλός προϋπολογισμός και το οφείλουμε αυτό να το δηλώσουμε. Καταρχάς, οι δηλώσεις αξιοπιστίας οι εθνικές δεν υποστηρίζονται από πολιτικά δεδομένα, δεν υπογράφονται από τον Υπουργό Οικονομίας ή από τον Πρωθυπουργό της κάθε χώρας, οπότε δεν γνωρίζουμε ποιος είναι υπεύθυνο για αυτές τις δηλώσεις εθνικής διαχείρισης των κοινωτικών ποσών. Αυτό λοιπόν δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, δημιουργεί παρανοήσεις και ατελείς εκθέσεις και παρουσιάσεις. Δεύτερον, σχετικά με τα ποσοστά λαθών, τα επίπεδα λαθών. Τα κράτη-μέλη πρέπει να επιστρέφουν τα χρήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν διαπιστώνονται τέτοια λάθη. Οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι πληρώνουν για τον κοινοτικό προϋπολογισμό και για μια ακόμη φορά οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι καλύπτουν τις ζημίες εισαγωγικά που δημιουργούνται, τα απρόβλητα δηλαδή αυτά ποσά, λόγω των λαθών, των απατών μερικές φορές που διαπιστώνονται στα πλαίσια της διαχείρισης των ευρωπαϊκών πιστώσεων. Θα ήθελα να ζητήσω να υπάρξει μια καλύτερη μορφή συνεργασίας ανάμεσα στο ελεγκτικό συνέδριο και τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια. Αν θέλουμε περισσότερα χρήματα στον κοινοτικό προϋπολογισμό, θα πρέπει να αποδείξουμε ότι τα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας είμαστε σε θέση να τα δαπανίσουμε με το σωστό τρόπο. Δυόμιση λεπτά Σε Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μπορούμε να μιλήσουμε για μία μείωση των λαθών σήμερα και αυτό το οφείλουμε στην επαγγελματικότητα και την αξιοπρέπεια του ελεγκτικού συνεδρίου το οποίο εκπροσωπεί ο κύριος Καλτέρα. Βέβαια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει βοηθήσει στη βελτίωση αυτή. Η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών είναι ιδιαίτερα προσεκτική σε σχέση με τη σωστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Θα πρέπει να βελτιώσουμε ακόμα τα πράγματα. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν ρυθμιστεί πλήρω, ιδιαίτερα σε ορισμένου τομεί όπω η γεωργία και η συνοχή. Έχουμε επίπεδα λαθών σε ορισμένου τομεί, τα οποία είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, όπω οι δημόσιε προμήθειε και οι υπερτιμολογήσει. Θα πρέπει να μειώσουμε καταρχάς το επίπεδο γραφειοκρατίας, να αποφύγουμε νομοθετικές ρυθμίσεις περιττές Θέλουμε λίγους κανόνες αλλά καθαρούς κανόνες. Έτσι θα απομακρύνουμε τις δυνατότητες, τον χώρο που δημιουργείται για λάθη αλλά και για απάτες και διαφθορά. Ένα άλλο θέμα που έχει αρκετά μεγάλη σημασία είναι να ενισχύσουμε τον ρόλο της ΟΛΑΦ, της υπηρεσίας που καταπολεμά τις απάτες και τη διαφθορά. Επίσης ένας άλλος τομέας, ε, τον οποίο δεν οφείλουμε να αγνοήσουμε βέβαια, είναι ο κίνδυνος ε, ε, να εμπλακεί στις διαδικασίες χορήγησης των ποσών αυτών σε χώρες όπως και στη δική μου άλλωστε το οργανωμένο έγκλημα. Απαιτείται λοιπόν μια καλή συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αποτρέψουμε τέτοιου είδους δυνατότητες. Πρέπει να πω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσει την αυτονομία της σε σχέση με τα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα ε, σε χώρες στις οποίες εδώ και λάθη διαπιστούνται πολύ σημαντικά λάθη, όχι μικρά λάθη και απάτες μερικές φορές, προς τις χώρες αυτές θα πρέπει να μπλοκάρονται τα ποσά και οι επιδοτήσεις για να αποφύγουμε τέτοιες επαναλήψεις ε, φαινομένων στο μέλλον. Νομίζω ότι η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξαρτηθεί από το επίπεδο διαφάνειας ε, το οποίο θα χαρακτηρίζει τη διαχείριση των κοινοτικών ποσών. Ευχαριστώ κύριε και Κύριος Βαντάλεν ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρόλο που το ελεγκτικό συνέδριο προβλέπει ε, ότι βελτιώθηκε ε, η κατάσταση ό,τι αφορά τις πληρωμές, δυστυχώς ε, δεν είναι πολύ θεωρητικά τα μηνύματα, γιατί υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις στη συνοχή, αλλά υπάρχουν ασφάλματα σε 40% των σχεδίων. Και 2 δισεκατομμύρια ουσιαστικά δεν δικαιολογούνται και να αχρεώστητα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγξει τον τρόπο με τον οποίο διαπράχθηκαν αυτά τα σφάλματα και να μειώσει αυτό το περιθώριο σφάλματος. Χθες ακούσαμε από το ελεκτικό συνέδριο ότι τα σφάλματα πολλές φορές οφείλονται στην περιπλοκότητα των διαδικασιών Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε απλούστερους και πιο διαφανείς μηχανισμούς. Αλλιώς ε, θα παραμείνει ένα πρόσιτο θέαμα για τους Ευρωπαίους πολίτες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Όμπερ Μάιερ. Κύριε Γκάιερ, θέλετε να παρέμβετε συζήτηση για το Catch αργότερα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχει δισεκατομμύρια ευρώ του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα, ένα λεπτό κύριε Οβερμαγερ. Ήθελα να δω. Η μπλε κάρτα ήταν η πραγματική παρέμβαση πλε κάρτα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, Είχα μια συμπραγματική ερώτηση στον συνάδελφο Φαντάλ. ήθελα να το ρωτήσω. Κύριε Φαντάλεν, δεχόσαστε μια ερώτηση, παρακαλώ. Ναι, ήθελα να ρωτήσω τον συνάδελφο Φαντάλεν κατά πόσον έλαβε υπόψη του ότι όσον αφορά τα υψηλά ποσοστά που ανέφερε, πρόκειται για τα ποσοστά των δειγματοληψιών. Δεν έχουμε 36% σφάλμα, ε, σφαλμένα κατά αχρεωσίους κατά Τα πραγματικά ε, στοιχεία είναι 5% και τα υψηλά ποσά δισεκατομμυρίων που αναφέρεται δεν είναι άλλα σωστά. Απάντηση. Κύριε, κύριε Πρόεδρε, το κατάλαβα, το έχω καταλάβει αυτό, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχουν δισεκατομμύρια που δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε πού πήγαν. Γι' αυτό ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγξει καλύτερα τα πράγματα και πιο διεξοδικά, προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση. Άλλωστε, ο ίδιο ο Επίτροπο είπε στην ομιλία του ότι ε, λαμβάνει αυτά τα, τα πορίσματα πολύ σοβαρά υπόψη και θα βαθύνει στι έρευνε. Ο κύριο Όπερ Μάγκερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 6 δισεκατομμύρια ευρώ του Ευρωπαϊκού Προπολισμού σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ηλεκτρικού συνεδρίου εξαφανίστηκαν το 2009. Γιατί, γιατί υπήρχε κακή διαχείριση, ε, ατασταλίες, απάτες και κακή διαχείριση. Παραδείγματος χάνει πολλές οικογένειες πήραν ε, διπλά εισοδήματα ε, και επιδόματα οικογένειας. Μια χώρα όπως η Ελλάδα η οποία είναι κύρια χώρα που απατά, παραδείγματος χάρη αν σκεφτώ πόσες επιφάνειες παίρνουν επιδοτήσεις για δασικές εκφράσεις κλπ. Δεν επιτρέπεται αυτό. Όπως είπε ο σας, από τις ελεγμένες ε, περιπτώσεις ε, από τις δειγματοληψίες είδαμε το 36% σφάλμα αυτό είναι απαράδεκτο. Θα πρέπει επιτέλους κύριε Επίτροπε κάτι να κάνετε. Δεν έχουμε χρήματα να τα πετάμε από το παράθυρο. Και επίσης θα ήθελα να συγχαρώ τους συνεργάτες του ηλεκτρικού συνεδρίου που είναι πραγματικά πολύ, ε, ε, πολύ ικανοί και θα πρέπει και στο μέλλον να συνδεστούν προς την ίδια κατεύθυνση. Ευχαριστώ κύριο Σόλμπρου και ένα, ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ. Η συζήτηση επί της ετήσιας έκθεσης απαιτεί κάποια ακρίβεια στην έκφραση απόψεων, γιατί πολύ ταυτόχρονα μιλούμε για τασταλίες, για σφάλματα, ακόμη και για απάτες. Η ετήσια έκθεση επισημαίνει ότι σε ό,τι αφορά το ποσοστό σφάλματος στην πολιτική συνοχή έχουμε σημαντική μείωση του σφάλματος και είναι κάτω από 5% αυτό το περιθώριο σφάλματος. Δεν μπορούμε λοιπόν να τα βάζουμε όλα στο ίδιο το τσουβάλι και να μιλούμε για ποσοστό σφάλματος 20, 30 ή και τα 100 γιατί έτσι αμαυρώνουμε την όλη εικόνα. Στην πολιτική συνοχή που είναι σίγουρα εξαιρετικά περίπλοκη και στηρίζεται στην κοινή διαχείριση μεταξύ και Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χωρών μερών υπάρχει βελτίωση. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα βελτιώσουμε αυτή την πολιτική που ίδια η δομή της είναι εξαιρετικά απαιτητική και πολυσύνθετη, περίπλοκη, αλλά έχει τεράστια προστιθέμενη αξία. Νομίζω ότι μπορούμε να εκφράσουμε την ε, ικανοποίησή μας για την θετική έκβαση. Βέβαια υπάρχει ένα αρκετά ανησυχητικό τμήμα στην έκθεση που λέει λαμβάνοντας ε, υπόψη τα προαναφερθέντα, το ελεκτικό συνέδριο θεωρεί ότι δεν μπορεί να δώσει θετική γνώμη σε ό,τι αφορά το επίπεδο σφαλμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΚΟΡΕΚ. Νομίζω ότι αυτή η διαπίστωση είναι πολύ σημαντική και θα είναι ουσιαστική για το μέλλον. Είναι Λίγες οι περιπτώσεις που δεν μπορεί το ελεκτικό συνέδριο να συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα αποτελέσματα όσο ό,τι αφορά το κόρεκ. Θα πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω αυτό το θέμα. Η κυρία Σχαλντεμόζη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ελεκτικό συνέδριο γιατί μας έδωσε πραγματικά ένα καλό μέσο εργασίας Όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των πόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε ότι ευτυχώ κινούμεθα προ τη σωστή κατεύθυνση, παρόλο που εξακολουθούν να παραμένουν προβλήματα. Το γεγονό ότι η κατεύθυνση είναι η σωστή Μα δίνει τη δυνατότητα να προγραμματίσουμε και το επόμενο βήμα. Να έχουμε δηλαδή επιτέλους ένα σωστό σύστημα ελέγχου για να έχουμε και λιγότερα σφάλματα. Αυτό δεν αρκεί όμως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξετάσουμε καλύτερα τη χρήση των χρημάτων αυτών κατά πόσον χρησιμοποιούνται σωστά όσον αφορά τη διαχείριση, τα κτίρια, το κόστος προσωπικού, κατά πόσον δηλαδή ε, ωφελούμεθα πραγματικά όπως πρέπει τα χρήματα αυτά, κατά πόσον πετυχαίνουμε το στόχο μας, θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή. Είναι και θέμα αποτελεσματικότητας και διαφάνειας. Πιστεύω ότι στο Κοινοβούλιο και στο Ελεκτρικό Συνέδριο και στην Επιτροπή θα πρέπει να το κάνουμε αυτό, να είμαστε πιο ανοιχτοί και να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Τσέσκοβα. Είναι η δεύτερη φορά όσο βρίσκομαι εδώ στο Κοινοβούλιο ενώ που συζητάμε την ετήσια έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ελεγκτές για την προσπάθεια την οποία έκαναν. Εκπλήσωμε ότι πράγματι υπάρχουν επίπεδα λαθών και απατών για ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των κοινοτικών πιστώσεων. Θα πρέπει να δούμε ποιος φταίει γι' αυτό. Η Επιτροπή φταίει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φταίνε τα κράτη-μέλη. Ποιος ακριβώς είναι ο υπεύθυνο. Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχει ανάγκη για βελτίωση της κατάστασης για να αποφύγουμε τέτοια λάθη στο μέλλον. Κύριος Ντόιτς, μισή λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, Το ελεγκτικό συνέδριο έπαιξε για μια ακόμη φορά το ρόλο του, ένα ρόλο εξαιρετικό σχετικά με την επιθεώρηση και τον έλεγχο του προϋπολογισμού και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2009. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Καλντέρα και όλους του τους ελεγκτές. Συμφωνώ με τους συναδέλφους οι οποίοι είπαν ότι η δήλωση αυτή δείχνει ξεκάθαρα ότι σχετικά με τη χρήση των κοινοτικών πιστώσεων τα πράγματα βαίνουν βελτιούμενα. Το ποσοστό των λαθών δηλαδή μικραίνει. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να καταλήξουμε νομίζω ήδη σε αυτή τη φάση σε ορισμένα συμπεράσματα. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν Ευρωπαϊκό Όργανο. Νομίζω ότι το, τα ποσοστά λάθους τα οποία εξακολουθούν να επιμένουν σήμερα ε, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι εκατομμύρια ευρώ χρησιμοποιούνται με απαράδεκτο τρόπο και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει ε, και δυνατότητα να διαπιστώσει κανείς ποινικά κολάσιμες ενέργειες. Συνεπώς θα πρέπει στις επόμενες δημοσιονομικές περιόδους να μας παρουσιάσει μία έκθεση το ελεγκτικό συνέδριο αναχώρα για να δούμε ποιες είναι οι χώρες οι οποίες σημειώνουν υψηλά επίπεδα μη κανονικών δαπανών. Τότε μόνο θα μπορέσουμε ουσιαστικά να μειώσουμε τα ποσοστά λάθους. Αγιάλα Σεντέρ. Ευχαριστώ. Για μία ακόμη φορά μπορούμε να εκφράσουμε την ευαρέσκειά μας για τις βελτιώσεις ε, που προσθέθηκαν χάρη στον επικοδομητικό διάλογο μεταξύ Ελεκτικού Συνεδρίου, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η φετινή έκθεση μας έδειξε ότι δεν θα πρέπει να επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας, αλλά να κρατήσουμε την επαγρύπνηση και την εγρήγορσή μας. Είναι σημαντική η πρόταση του κ. Καλδέρα για το μέλλον σε ό,τι αφορά τη βελτίωση του συντονισμού και τη συνεργασία για να βελτιώσουμε σημαντικέ πτυχέ του δημοσιονομικού κανονισμού, έχοντα υπόψη και το μέλλον και τι ε, μελλοντικέ νομοθετικέ προτάσει, τι οποίε ε, χάρη στη συνεργασία μα θα έχουμε και βελτίωση. Εγώ θα είμαι ιδιαίτερη ιδιαίτερα προσεκτική για τις λειτουργικές ε, δαπάνες του Συμβουλίου, ιδιαίτερα για το σύστημα ΣΕΖΑΜ. Εκεί αναφέρεται ειδικά η ανάγκη βελτίωσης σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις για το, στον προϋπολογισμό του Συμβουλίου. Επίσης, ε, με μονομένες πτυχές όπως ε, το θέμα του διαμεσολαβητή, της προστασίας των δεδομένων, φαίνονται κάπως υποβαθμισμένα αυτά τα σημεία. Επίσης, δόθηκαν κάποιες πληροφορίες ε, για κάποιες υποθέσεις που διαβάστηκαν στην ΟΛΑΦ από την ΟΚΕ. Και θα ήθελα να ρωτήσω γιατί αυξήθηκε τόσο πολύ το προσωπικό της Επιτροπής Περιφερειών τα τελευταία χρόνια. Η κυρία Ιβάνοβα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα συμπεράσματα του ελεγκτικού συνεδρίου για το 2009 δεν διαφοροποιούνται ε, με τα αντίστοιχα συμπεράσματα των προηγούμενων ετών. Ελάχιστα τουλάχιστον διαφοροποιούνται. Έχουμε επανειλημμένα στο Κοινοβούλιο αυτό ζητήσει να ληφθούν νέα μέτρα, ιδιαίτερα σε τομείς τους οποίους διαπιστώνονται υψηλά επίπεδα δυσλειτουργιών. Θα θέλαμε να απαλλαγούμε από τις δυσλειτουργίες αυτές. Για το 2008 υπήρξε μία βελτίωση και στον τομέα της πολιτικής συνοχής. Παρ' όλα αυτά η κατάσταση ε, δεν φαίνεται να βαίνει συστηματικά ε, βελτιούμενη. Μπορεί τα πράγματα να αλλάξουν ανάλογα με τις συνθήκες οι οποίες ε, επικρατούν σε κάθε κράτος μέλος. Υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες και σε άλλες πολιτικές όπως η διεύρυνση, η βοήθεια για την ανάπτυξη, η ενέργεια, οι μεταφορές, η εκπαίδευση και η έρευνα. Ως εκ τούτου θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει περισσότερες προσπάθειες και να συνεργαστεί με την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Προϋπολογισμού για να βελτιωθεί η χρήση των κοινοτικών πιστώσεων. Ο κύριος Γκάιερ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξωτιμή κύριε Πρόεδρε Καλτέρα, εξωτιμή κύριε Επίτροπε. Η ε, η πολιτική συνοχή είναι ο μεγάλο ασθενή Πέρσι ήταν στην εντατική, σήμερα είναι σε ανάρρωση, αλλά ακόμα δεν είναι υγιή απόλυτα και υπάρχει ο κίνδυνος ε, να ξανακαταρρεύσει. Το 5% ήταν ασφαλμένες καταβολές, το 3% δεν θα πρέπει να έχουν καταβληθεί, ένα συνολικό ποσό 700 εκατομμυρίων ευρώ, ένα μεγάλο ποσοστό των αχρεωστήτως κατεβληθέντων ποσών είναι ευθύνη των κρατών μελών. Εδώ γίνονται τα σφάλματα. Και αυτό παρόλο το συστήματα ελέγχου που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και έχουν εγκαθιδρυθεί από την Κομισιόν, θα πρέπει νομίζω να ξανεκταστούν τα συστήματα αυτά ελέγχου. Στη χώρα μου, τη Γερμανία, οι δειγματοληψίες απόδειξαν ότι όλα τα συστήματα ελέγχου που ε, εξετάστηκαν ήταν μόνο μερικώς αποτελεσματικά η ευθύνη υπάρχει στα χέρια της Κομισιόν. Δηλαδή υπάρχει εδώ μια αντίφαση. Τα σφάλματα είναι στα κράτη-μέλη και η ευθύνη είναι στην Κομισιόν. Μπορούμε να το συζητήσουμε στις ε, ε, χώρες μας. Αλλά πολιτικά είναι θέμα της Κομισιόν να το επιβάλλει στα κράτη-μέλη. Κύριε Σέμετα, είστε πιο αυστηρός. Θα είμαστε στο πλευρό σας. Ευχαριστώ. Ε, το λόγο έχει ο κύριος Βανίλ Στερόι για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε του Ελεκτικού Συνεδρίου, κύριε Επίτροπε, κυρίε και κύριοι, είμαι ο συντονιστή του ΕΛΚ για την περιφερειακή πολιτική. Το ποσοστό σφάλματος ε, για την πολιτική συνοχή φαίνεται ότι έχει μειωθεί. Είναι πολύ θετικό αυτό. Βέβαια έχουμε τον νέο κανονισμό και τα σχέδια δράσης που ζητούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που ξεκίνησε η προηγούμενη Επιτροπή. Διαπιστώνουμε όμως ότι πολλά από τα σφάλματα αυτά σχετίζονται με προκηρύξεις διαγωνισμών, με δημόσιες προμήθειες, με μεταφορά, με ενσωμάτωση του κοινοτικού δικαίου στην εσωτερική ένωμη τάξη, με την εκτέλεση των διατάξεων αυτών. Η ελληπής αυτή εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου αυξάνει πολλές φορές το ποσοστό σφάλματος. Θα πρέπει να ασκήσουμε κάποια πίεση στα κράτη-μέλη ή να τα υποστηρίξουμε στους δημόσιους αυτούς διαγωνισμούς. Πραγματοποίησα επίσκεψη στην Ρουμανία και είδαμε ότι υπάρχουν προβλήματα εκεί. Γι' αυτό θα πρέπει να εργαστούμε άοκνα για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Εγώ είμαι υπέρ των εθνικών, λογαριασμών, ε, ε, εθνικών δηλώσεων διαχείρισης που θα υπογράφουν οι Υπουργοί Οικονομικών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βόγκαν για ένα λεπτό. Uh, uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να είμαι όσο πιο θετικός μπορώ σε σχέση με αυτή την έκθεση. Πρέπει να χρησιμοποιούμε τις εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου για να βελτιώνουμε τα πράγματα, να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και υπάρχουν παραδείγματα όπου κάτι τέτοιο έχει πράγματι διαπιστωθεί και έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Στη Γεωργία σαν παράδειγμα οι συνεχείς αλλαγές των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημιουργούν δυσκολίες στους ε, γεωργούς και στα κράτη-μέλη. Αυτό μου λένε συνεχώς στην Ουαλία. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν να αλλάξει την ομοθεσία η οποία περιγράφει και ορίζει τους σε ενέργεια ε, γεωργούς στο Ηνωμένο Βασίλειο και συνολικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει λοιπόν χώρος εδώ για απλούστευση των διαδικασιών έτσι ώστε στην Ευρώπη να ελέγχουμε σωστά τα χρήματα τα οποία δαπανούμε για συγκεκριμένο όφελος των πολιτών και των κοινοτήτων μας. Περνάω στη διαδικασία Catch the Eye. Το λόγο έχει κύριος Γκζίμπ για ένα λεπτό. Φαντάζομαι αυτό εννοούσε. Ο κύριος Γκζίμπ. Ευχαριστώ η παρουσίαση αυτή της αιτήσιας έκθεσης του Ελεκτικού Συνεδρίου μας ε, δίνει πολύ σημαντικές ε, γνώσεις και μπορούμε να συγκρίνουμε την κατάσταση με το παρελθόν και να προγραμματίσουμε τις δράσεις μας για το μέλλον. Ε, όσο πιο εύκολε είναι οι διαδικασίε, όσο πιο πλούστερες είναι οι διαδικασίε, τόσο μειώνεται και το ποσοστό ε, σημαντικών σφαλμάτων. Όσο πιο περίπλοκες είναι οι πολιτικέ, τόσο ε, πιο ουσιώδη σφάλματα έχουμε και τόσο περισσότερες ατασταλίες παρατηρούμε. Η πολιτική συνοχή είναι εξαιρετικά σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό φυσικά διαπιστώνουμε ότι και η κοινή γεωρική πολιτική ε, είναι περίπλοκη και παρατηρούμε σημαντικό ποσοστό σφάλματος, αλλά ίσως οφείλεται και πάλι στην περιπλοκότητα των διαδικασιών. Είναι σημαντική η συνεργασία μεταξύ των ελεκτικών οργάνων, αλλά είναι σημαντική και η συνεργασία μεταξύ των ε, κοινοβουλίων και του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού. Οι πληροφορίες αυτές ήταν πολύ χρήσιμες και διαπιστώσαμε ότι ήταν ε, πολύ θετική η υποδοχή της έκθεσης του Ελεκτικού Συνεδρίου και από τους Εθνικούς Βουλευτές. Κυρία Κάλεμπαχ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ το Ελεκτικό Συνέδριο. Νομίζω ότι η έκθεση δείχνει πραγματικά εντυπωσιακά ότι οι έλεγχοι όσο πάει και βελτιώνονται και δεν τρομάζω πάντα από τα ποσοστά ασφάλματο, γιατί νομίζω ότι και ο έλεγχο του λογαριασμού είναι μια διαδικασία που μαθαίνεται ε, καθοδόν και είναι καλό που όσο πάει και περισσότερα ασφάλματα βρίσκουμε. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε από κοινού για να αποφύγουμε τα ασφάλματα αυτά στο μέλλον και ε, χαίρομαι ε, όπου μπορώ να πιστεύω την προσοχή σας στην πέμπτη έκθεση ε, συνοχής που παρουσιάστηκε χθε γιατί η Κομισιόν καλεί τους πάντες να τοποθετούν πάνω στο θέμα αυτό. Εδώ έχουμε μια δυνατότητα ε, να θέσουμε τους όρους και για το μέλλον, τόσο ώστε αφενός οι ενισχύσεις στον ένα τομέα να είναι πιο εύκολες, στο να μειωθεί δηλαδή η γραφειοκρατία στο μέλλον και από την άλλη μεριά να έχουμε καθαρό έλεγχο για τη χρήση των ε, φορολογικών εισόδων και καλώ όλους να εκλε... ακολουθήσουν με αυτή όπως το κάνουμε και μέσα στο κοινοβούλιο. Ευχαριστώ λέει πρόεδρος. Δεν βλέπω κανένα άλλο να ζητάει κάτι. Ε, ε. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στον Επίτροπο Σεμέτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η συζήτηση που προηγήθηκε δείχνει ότι έχει υπάρξει περαιτέρω πρόοδο στην διαχείριση του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού για το 2009. Αυτό ε, μας επιτρέπει να θεωρήσουμε αξιόπιστες ε, τις, ε, τα στοιχεία αυτά και να θεωρήσουμε επίσης σωστά τα μέτρα τα οποία πήραμε για την βελτίωση των προγραμμάτων της ίδιας δημοσιονομικής περίοδου. Το συνέδριο βέβαια εντοπίζει και ορισμένους τομείς τους οποίους απαιτείται να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος και αναφέρομαι και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και στους ε, οικονομικούς εταίρους μας, τα κράτη-μέλη δηλαδή, που θα πρέπει ε, να ε, ενισχύσουν ακόμα καλύτερα τους τρόπους ελέγχου. Άκουσα εδώ διάφορα από τους ομιλητές για τα θέματα των κυρώσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβάλλει κυρώσεις και με μεγάλη αυστηρότητα. Είμαστε στη διαδικασία διακοπής 40 ε, προγραμμάτων στον τομέα της συνοχής, συνολικά 1 δις 750 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Και αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι ο αριθμός των ενεργειών το 2010 σε σχέση με την επιβολή κυρώσεων έχει διπλασιαστεί σε σχέση με τις αντίστοιχες περιπτώσεις του 2008 ή 2009. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα την απόφαση πήραμε μια, πήραμε μια απόφαση να ανακτήσουμε ποσά τα οποία ξεπερνούν σχεδόν τα 600 εκατομμύρια ευρώ. Εφαρμόζουμε λοιπόν το σύστημα των κυρώσεων αυστηρότατα και θα συνεχίσουμε να το εφαρμόζουμε και στο μέλλον. Από την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου φαίνεται ότι το επίπεδο ανακτήσεων αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια και το 2009 έφτασε τα 3 δις 300 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς, εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια την οποία κάνουμε, επιβάλλοντας ανάμεσα σε άλλα και κυρώσεις όπου αυτό χρειάζεται. Η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου λοιπόν και η διαδικασία απαλλαγής που μόλις ξεκινά όχι μόνο θα διορθώσει τις αδυναμίες του υπάρχοντος προγράμματος αλλά θα δημιουργήσει και βελτιώσεις και στις μελλοντικέ χρήσεις. Και εδώ έχουμε περαιτέρω μέτρα να λάβουμε στον τομέα της απλούστευσης της νομοθεσίας, των κανόνων προμηθειών. Είναι αλήθεια ότι πολύ μεγάλα ποσοστά λαθών οφείλονται ε, στην παραβίαση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και ιδιαίτερα στον τομέα των δημοσίων προμηθειών πρέπει να, να καταλήξουμε στα κατάλληλα συμπεράσματα. Λοιπόν, θα εφαρμόσουμε τις συστάσεις του συνεδρίου και ελπίζουμε και η διαδικασία απαλλαγής να είναι εξίσου κακοφόρα. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση να δώσω το λόγο στον ε, πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου, τον κύριο Σίλβα Καλντέρα. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Αξιότιμη Ευρωβουλευτέ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους Ευρωβουλευτές για τα πολύ ευγενικά του σχόλια και τις φιλοφρονίες τους προς το ελεκτικό συνέδριο. Προσπαθούμε στο ελεγκτικό συνέδριο να εφαρμόσουμε τις ε, πλέον ποιοτικέ και υψηλέ προδιαγραφές ελέγχου εφάμιλες με τις υψηλέ ελεκτικές προδιαγραφές όλων των ε, διεθνών οργανισμών. Θα ήθελα να σας δώσω δύο παραδείγματα από την ετήσια έκθεση του 2009 για να δείτε τι κάνουμε προκειμένου να ανταποκριθούμε στο έτοιμά σας για καλύτερη ενημέρωση. Πρέπει σε μια συνολική αξιολόγηση της κατάστασης και για πρώτη φορά δίνουμε μια σφαιρική εικόνα της κατάστασης και μάλιστα διαπιστώνουμε μια βελτίωση τα τελευταία χρόνια. Και για το σύνολο του κοινοτικού προπολογισμού το ποσοστό σφάλματος μειώνεται. Και μάλιστα ιδιαίτερα στον τομέα της συνοχής σας δίνουμε πολύ περισσότερες πληροφορίες από ότι πέρυσι. Γιατί στην περσινή ετήσια έκθεση είπαμε ότι τουλάχιστον 11% των κονδυλίων δεν θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί. Ενώ φέτος μπορούμε να δηλώσουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα το ποσοστό σφάλματος είναι λίγο πάνω από το 5%. Κάτι που δεν μπορούσαμε να ισχυριστούμε πέρυσι και λέμε ότι τουλάχιστον 3% των κονδυλίων δεν θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί. Αυτό δεν είναι και το μέτρο της πρόοδου που διαπιστώσαμε στη φετινή μας έκθεση. Έχουμε σημειώσει πρόοδο λοιπόν. Για ποιο λόγο. Δεν ε, επινοούμε εμείς αυτά τα στοιχεία. Δεν θέλουμε να είμαστε ούτε επικείς ούτε αύριο απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Το ελεκτικό συνέδριο είναι ανεξάρτητο φορέας, ανεξάρτητο οργανισμός, κατοχυρώνεται από τη συνθήκη και στηρίζει τα πορίσματά του σε τεκμήρια, σε αποδείξει. Και σε αυτές τι αποδείξεις στηρίζουμε την έκθεσή μα. Αυτή είναι η υποχρέωσή μα. Να σα βοηθήσουμε για τη διαδικασία τη απαλλαγή. Είμαστε λοιπόν πρόθυμοι να σας βοηθήσουμε στο έργο σας. Και ο βασικός λόγος γι' αυτό, όπως είπαμε και στην ετήσια μας έκθεση, είναι ότι τα συστήματα για τη διαχείριση των προγραμμάτων για την περίοδο 2007-2013 έχουν καλύτερες επιδόσεις πια. Ένας άλλος λόγος είναι ότι η καταβολή των κονδυλίων για την περίοδο προγραμματισμού είναι μόνο 25%. Οπότε η δημοσιονομική εκτέλεση για την περίοδο αυτή, κατά τη γνώμη μας, είναι χαμηλή, χαμηλότερη από ό,τι αναμενόταν. Ο συνδυασμός λοιπόν αυτών των δύο παραγόντων, της απόδοσης του συστήματος, βελτιωμένης απόδοσης του συστήματος και χαμηλότερης εκτέλεσης, άρα λιγότερων πληρωμών, οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση. Γι' αυτό είπαμε ότι θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Γιατί θέλουμε ένα σύστημα που θα είναι αποδοτικό και στις 27 χώρες μέλη. Και θέλουμε στο μέλλον τα κονδύλια να δαπανώνται, να απορροφώνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να εκταμιεύονται σωστά. Γι' αυτό είπαμε ότι επειδή αυτή η κατάσταση δεν ισχύει ακόμη, να είμαστε επιφυλακτικοί. Φυσικά είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού για τη διαδικασία της απαλλαγής. Οι τα μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου θα σας βοηθήσουν στη διαδικασία απαλλαγής χορηγώντας σας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Αλλά και με τις ειδικέ μας εκθέσεις σας βοηθούμε. Υπάρχουν πολλές εκθέσεις ειδικέ με βάση τους ελέγχους που πραγματοποιήσαμε και νομίζω ότι χρησιμοποιούνται γιατί είναι, περιλαμβάνουν πολύτιμες πληροφορίες και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά τις ευθύνε για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, ε, κύριοι υπεύθυνοι για την εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συνθήκη της Λισαβόνας όμως προβλέπει εκτέλεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Οπότε μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι σήμερα έχουμε μία μοναδική ευκαιρία για να προβούμε σε μια καλύτερη διαχείριση του κοινοτικού προπολογισμού. Έχουμε ένα νέο δημοσιονομικό κανονισμό που εξετάζεται αυτή τη στιγμή και θα εγκριθεί σε το χρόνο και αυτό θα είναι ο βασικός προσανατολισμός που θα μας οδηγήσει και στο μέλλον προκειμένου να έχουμε βελτίωση, πρόοδο, αν θέλουμε να έχουμε απλούστερους κανόνες πιο αποτελεσματικά συστήματα, με καλύτερη απόδοση κόστους ωφέλους. Αυτά θέλουμε και αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία για να προωθήσουμε όλες αυτές τις αλλαγές. Και θα είναι επιτάπητος η αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού και του χρόνου. Ε, λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση που χρήζει σημαντικών αποφάσεων για τη βελτίωση στο μέλλον. Και αν μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε ελεκτικό συνέδριο, θα σας έλεγα να αξιοποιήσετε τις συστάσεις μας, γιατί στην έκθεσή μας περιλαμβάνονται συστάσεις για τις βασικές προκλήσεις και τους τρόπους βελτίωσης της χρηματοοικονομικής, της δημοσιονομικής διαχείρισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την περίοδο μετά το 2013. Θα πρέπει να διαρωτηθούμε τα προγράμματα και τα χρηματοδοτικά συστήματα θα προσφέρουν προστιθεμένη αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε συστήματα και προγράμματα που είναι σαφή, απλά, με στόχους ε, κατανοητούς και ρεαλιστικούς. Και η λογοδοσία, οι κανόνες λογοδοσίας και η υπευθυνότητα είναι σαφείς, γιατί μερικές φορές ε, ε, πολλοί αποποιούνται των ευθυνών τους και κανένα δεν θέλει να αναλάβει να υπομισθεί τι ευθύνε, ότι η Επιτροπή, τα κράτη-μέλη. Το ελεκτικό συνέδριο βρίσκεται εδώ για να σα βοηθήσει προκειμένου να υλοποιήσουμε όλε αυτέ τι προκλήσει. Ευχαριστώ. Κλείνει συνεπώ η συζήτηση εδώ. Περνάμε τώρα στην έκθεση Van Brent για την τροποποίηση του κανονισμού 663 του 2009.